διαβάσω τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση στα πρόσωπα και τους φορείς τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στα ψηφίσματα. Η παρούσα σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται. Η συνεδρίαση έληξε.